Uh, uh, Ωραία, μπορούμε να ξεκινήσουμε την δημοσία Θα μιλήσω σου ειδικά. Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ για να καταλαβαίνετε και τι λέω. Καλωσορίσατε όλοι στην Επιτροπή τη δική μας σε μια ακρόαση που έχουμε ε, συζητάμε για καλύτερους μηχανισμούς για ε, θεσμική και ε, δικαστική ισότητα άνδρες-γυναίκες. Έχουμε κάποιες γνώσεις και εμπειρία και χαίρομαι που έχουν έρθει εδώ πέρα οι καλεσμένοι μας σήμερα. Μας ικανοποιεί αυτό. Είσαστε εμπειρογνώμονες και όταν μιλάει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα λέμε ότι πρέπει να πιάσουμε ένα υψηλό ελάχιστο επίπεδο. Δημιουργούνται πολλοί συμβιβασμοί για να πετύχουμε αυτό το επίπεδο στο οποίο θα συμφωνήσουν όλοι. Εδώ καταλήγουμε συχνά σε πράγματα τα οποία αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα. Η ισότητα είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Ε, τα, τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό θα ήταν καλό να έχουμε σαν ένα στόχο να πετύχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο δικός μας, θα λέγαμε, ο ο αστέρας ο οποίος μας οδηγεί. Και μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλο, από τις κοινότητές μας και πραγματικά ο στόχος μας θα έπρεπε να είναι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Έτσι θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα έχει και καλύτερη, το καλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Λοιπόν, εγώ είμαι υποστηρικτής, μεγάλος υποστηρικτής αυτού που λέμε best practices. Εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό όταν κανείς συναντάει άλλους ανθρώπους με άλλες ιδέες και έχουν διακριθεί σε αυτό να μπορέμε να τα δούμε αυτό και να μάθουμε για αυτό το πράγμα σε τοπικό, ε, κοινωτικό επίπεδο. Να μπορέσουμε να συζητούμε ο ένας με τον άλλον. Ίσως, ενδεχομένως, να μην μπορεί κανείς να υιοθετήσει μια πολύ καλή ε, εφαρμογή σε μια χώρα και να την περάσει στη δική του. Ίσως αυτό να μην είναι πάντοτε δυνατό. Αλλά πιστεύω ε, αυτό μπορεί να εμπνέει κάποιον οι ιδέες εμπνέεται κανείς από προτάσεις και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θετικά πράγματα. Γι' αυτό χαίρομαι, χαιρόμαστε μάλλον που είμαστε εδώ πέρα, που έχουμε τους καλεσμένους Δεν θα μιλήσω παραπάνω, Είμαστε ήδη λίγο ελαφρώς καθυστερημένοι. Λοιπόν, ξέρετε, ε, για ένα Σκανδιναβό αυτό το πράγμα, πέντε λεφτά καθυστέρηση είναι μεγάλη. Λοιπόν, αμέσως θα δώσω το λόγο στον, στην αντιπρόεδρο Ελίζα Μόρι Αρτιέ, η οποία θα είναι αντιπρόεδρος για αυτήν εδώ την ε, σημερινή ε, συζήτηση. Χαίρομαι που η Ελίζαμπετ θα αναλάβει να σήμερα το συντονισμό θα έλεγα αυτής της συνάντησης. Έλα θα εδώ στη θέση μου. Bonjour, mais... Καλησπέρα σας. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Σόρεν, τον πρόεδρό μας, της Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Πολιτών, τον κύριο Γκούφτασο δηλαδή, να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανη που ένας άντρας έχει αναλάβει την Προεδρία αυτής της Επιτροπής, ώστε να επιδιώξουμε τη φιλοδοξία αυτή που εδώ και δύο χρόνια προσπαθούμε να οργανώσουμε, δηλαδή να έχουμε μια ακρόαση για την ρήτρα της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας. Πρόεδρε, είναι ένα πολύ καλό μήνυμα αυτό ανοιχτού πνεύματος και κινητοποίησης για τον στόχο μας έναν στόχο για τον οποίο όλοι ενδιαφερόμαστε και κοινοτοποιούμαστε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που βρίσκονται ήδη εδώ. Θα έρθουν και άλλοι φαντάζομαι. Ευχαριστώ λοιπόν όσες και όσους έχουν αναλάβει δράση, προσήλθαν για να συμμετάσχουν σε αυτή την ακρόαση. Η ακρόαση αυτή μας θέτει ενώπιον ενός διτού προβλήματος. Το πρώτο σκέλος είναι αυτό του να οικοδομήσουμε από κοινού την ισότητα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Επίπεδα που αφορούν την καθημερινή, τον καθημερινό μας βίο. Η φιλοδοξία αυτή έχει λάβει κατεπήγοντα χαρακτήρα επειδή διανύουμε μια περίοδο κρίσης περίοδο που κάνει σε σημαντικό βαθμό ακόμα πιο αμφίβολη και ευάλωτη την ισότητα μεταξύ των πολιτών. ισότητα που δύσκολα επιτυγχάνεται αλλά δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από την κρίση. Κατά την άποψή μου ε, αυτό το επιχείρημα πρέπει όλους να μας οδηγήσει στη δράση και μας αφορά όλους. Ξέρετε ότι εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας για τις γυναίκες λοιπόν και την απασχόληση στην περίοδο της κρίσης Πρέπει να ευχαριστήσω κατά πρώτον την ε, Μαρία Γκαμπριέλ, συντονίστρια του ΕΛΚ, που μου ανέθεσε την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Όμως βλέπουμε ότι εδώ έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη στους ώμους μας για αυτό το πεδίο δράσης. Και το δεύτερο σκέλος για το οποίο οφείλουμε να αναλάβουμε δράση είναι ότι για έναν τέτοιο στόχο τίποτε δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Το σύνολο των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, ευρωπαϊκό, εθνικό, όπως το είπατε και εσείς πρόεδρε, και τοπικό, οι ενώσεις, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλα πρέπει να συνδυαστούν. Ο μοχλός, η κινητήριος δύναμη που θα μας οδηγήσει να υλοποιήσουμε, να επιδιώξουμε την ισότητα των πολιτών, όλα θα πρέπει να τα αξιοποιούμε. Έτσι τίθεται το θέμα της διάρθρωσης μεταξύ ευρωπαϊκού δικαίου και εθνικού δικαίου. Εθνικών μάλλον δικαίων. Έτσι λοιπόν, και αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι που μου αρέσει τόσο σε ένα θέμα όπως το σημερινό, έτσι πρέπει όχι μόνο να εργαστούμε για την, και να κοπιάσουμε για την ισότητα μεταξύ των πολιτών, αλλά έχουμε ένα πεδίο δράσης πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή να συνδυάσουμε το ζών έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό των κρατών μελών. Νομίζω ότι είναι μια από τις δυσκολίες του έργου που έχουμε αναλάβει αλλά είναι και μια επιπλέον ευχαρίστηση. Να κινητοποιήσουμε την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας, παίρνοντας αφορμή από ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, πολύ χειροπιαστό. Ισότητα ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερο τις εμπειρογνώμονες που μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας. Έχουμε μια πολύ ωραία ομάδα εμπειρογνωμόνων και πιστεύω ότι θα σας ευχαριστήσει όλους η παρουσία τους. Καταρχάς θα ακούσουμε την Σεβρίν Ντυπανή. Είναι στρατευμένη η Σεβρίν και πολύ δραστήρια είναι μία από τις συγγραφείς του βιβλίου με θέμα ακριβώς της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας, τη ρήτρα για την πλέον ευνοημένη Ευρωπαία. Είστε ειδική νομικός ε, σύμβουλος και εξειδικευμένη στο ευρωπαϊκό δίκαιο και χάρη σε εσά, στις δικές σας μελέτες και τις έρευνες έχετε ζήσει στην ε, Αγγλία, στην Ιταλία στη Γαλλία. Έχετε βοηθήσει όλες τις Ευρωπαίες, έχετε δημιουργήσει μια... έχετε καταλήξει σε μια επισκόπηση του πώς έχει η κατάσταση στην Ευρώπη και έχετε ασχοληθεί και με το πώς διορθώνεται το έργο των θεσμικών οργάνων μεταξύ τους σε εθνικό επίπεδο, λόγω χάρη με το έργο του Γαλλικού Κοινοβουλίου ασχοληθήκατε, αλλά και και με εμπορικά επιμελητήρια όπως αυτό για, τους, για τη βιοτεχνία. Η κυρία Ντυπανή λοιπόν θα μας μιλήσει για το έργο της Ένωσης. Ε, επιλέγουμε το δίκαιο των γυναικών και μετά θα έχουμε την εισήγηση του Ζαν ο οποίος είναι καθηγητής, ε, επίκουρος καθηγητής στο Παρίντο Φιν και κυβερνητικός ε, σύμβουλος. Ξέρω ότι είστε πολύ άσχολος και είναι πολύτιμος ο χρόνος σας. Όμως και εσείς διαθέτετε ιδιαίτερες γνώσεις για το δημόσιο δίκαιο και το κοινοτικό δίκαιο στα θέματα αυτά και τη διάρθρωση ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου πείρα και οι δικές σας γνώσεις σε αυτόν τον τομέα θα μας είναι πολύτιμες. Είστε συγγραφέας ε, πολλαπλών ε, πονημάτων για το θέμα αυτό και θα είναι τιμή μας να σας ακούσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε να, φω... να μας φωτίσετε με τις ιδιαίτερες γνώσεις σας. Και έπειτα θα έχουμε την τρίτη μας εμπειρογνωμονά, την κυρία Μίκε Βερλό. Με συγχωρείτε, πρέπει να προφέρω άσχημα το όνομά σας. Αλλά είναι πραγματικά χαρά μου να σας ε, υποδέχομαι εδώ. Είστε ε, καθηγητής συγκριτικής πολιτικής, συγκριτικών πολιτικών επιστημών σε θέματα ισότητας στο Πανεπιστήμιο του Νουμέκ και έχετε μεγάλη πείρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξατε σύμβουλος πολλών ευρωπαϊκών ε, κυβερνήσεων και έχετε αναλάβει διαφορετικά πόστα σε πολλές ευκαιρίες, οπότε η δική σας γνώση μας είναι επίσης πολύτιμη. Σας ευχαριστούμε και εσάς λοιπόν, κυρία καθηγήτρια, που μπορείτε να μας παρουσιάσετε το απόσταγμα των μελετών και των ερευνών σας. Χωρίς, περαιτέρω, χωρίς να χρονοτεπίσω περαιτέρω, νομίζω ότι κατεπήγε να σας αφήσω το λόγο και ε, να ακούσουμε εσάς πρώτα, κυρία Ντυπανή. Καλημέρα και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και επίση τον πρόεδρο τη Επιτροπή, τον κύριο Κουστέρσον που μα έδωσε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σήμερα στην Επιτροπή σα. είμαστε ιδιαίτερων ευγνώμονε και θα ήθελα να σα μεταφέρω και εκ μέρου τη κυρία Χαλινή, που είναι πρόεδρο τη οργάνωση μα Σοζή Λεκό Δεφάμ. Δυστυχώ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί, γιατί ε, εκπροσωπεί την οργάνωση μα στην Αλγερία. Παρ' όλα αυτά, ε, σας ευχαριστούμε για την ε, πρόσκληση και ε, σας, ευχαριστώ και, σας ευχαριστώ και εκ μέρους της κυρίας Χαλίμη. Εδώ και πέντε χρόνια έχουμε επαφές και συνεργασία με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των διοφύρλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη και, και, και επικοδομητική συνεργασία είχαμε μεμονωμένες ε, επαφές και συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και ορίστε λοιπόν γιατί είμαστε ιδιαίτερος ευτυχείς που θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε άμεσα στα μέλη της Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα, μια μικρή παρουσίαση της ε, οργάνωσής μας και του ιστορικού για όσους ε, δεν γνωρίζουν εις βάθος πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 1971 από την Simone de Beauvoir, τον Ζιζέλ Χαλιμή και τον Ζακ Μονό. Είναι μια οργάνωση ανεξάρτητη από τα πολιτικά κόμματα και προσπαθεί να προωθήσει την ανάλυση των δικαιωμάτων και της ισότητας των δύο φύλων. δημιουργία της οργάνωσης ακολούθησε την ε, δίκη της, ε, του Μπομπινί, στην οποία το θύμα ενός βιασμού έκανε έκτρωση. Εκείνη την εποχή αυτό ήταν παράνομο στη Γαλλία. Ακολούθησε δίκη, στην οποία καταδικάστηκε και αυτό προκάλεσε μια δημόσια συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών. Μέσα από αυτήν την ε, δημόσια συζήτηση δημιουργήθηκε και η οργάνωσή μας. Μετά αυτήν την δίκη ε, υιοθετήθηκε ένας, ε, ο νόμος Βέιλ, στην Σιμών Βέιλ, στη Γαλλία, η οποίο έδινε την δυνατότητα στις γυναίκες που είχαν υποστεί βιασμό να νομίμως να κάνουν έκτρωση. Η οργάνωσή μας κατόπιν έχει ε, ε, ασχοληθεί με τα ζητήματα της εκπροσώπησης των γυναικών στην πολιτική ζωή, στέλνοντας τις, τους πρώτους παρατηρητές για ζητήματα ισότητας και δημιουργώντας το παρατηρητήριο για ζητήματα ισότητας. κάτι που οδήγησε και στην αναθεώρηση του Γαλλικού Συντάγματο και την υιοθέτηση, την θεσμοθέτηση μάλλον τη ε, ισότητα των δύο φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή. Έρχομαι στο ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα, τη ρήτρα της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας. είναι μια έννοια η οποία ξεκίνησε από το 1979. Και γιατί αυτό. Τότε ήταν η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέχθηκε με καθολική ψηφοφορία. Οι φεμινίστριες λοιπόν εκείνη την εποχή έθεσαν το ζήτημα του τι σε τι βοηθά, σε τι βοηθά αυτή η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ίδιας τη γυναίκες. Οι ιδέες που συνέλαβε η, η πρώτη πρόεδρος της οργάνωσής μας εκείνη την εποχή έλαβαν σάρκα και οστά πολύ αργότερα. δημιουργήθηκε μια επιτροπή από εθελοντές, από εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων, νομικούς, ε, αγωνίστρες για τα δικαιώματα των γυναικών, η οποία είχε ως στόχο να κάνει έναν απολογισμό και να συλλέξει τεκμηρίωση όλης της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των γυναικών. Και εμείς συνεχίσαμε αυτήν την διαδικασία μελέτης, η οποία ήταν αρκετά περίπλοκη, υπήρχε το ζήτημα της μετάφρασης, υπήρχε το θέμα της επαφής με τις ε, πρεσβείες προκειμένου να συλλέξουμε τη σχετική νομοθεσία και καταλήξαμε σε μια σύνθεση, μια συνολική ε, εικόνα στην οποία έχουμε ε, καταγράψει τον ισχύουσα εθνική νομοθεσία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε, ό,τι, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τι γυναίκε, και σε καθένα από αυτά τα ζητήματα έχουμε επιλέξει τι ρήτρε, τι διατάξει, τι πλέον ευνοϊκές για τι γυναίκε. Στα ζητήματα τη ενδοοικογενειακή βία, τη βία κατά των γυναικών, στον, στον τομέα τη αγορά εργασία, στην ισότητα στην εκπροσώπηση, στην εκπροσώπηση στις πολιτικές αποφάσεις, αλλά επίση και στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, καθώ επίση και το οικογενειακό δίκαιο τις σχέσεις τέκνου γονέα, ζητήματα εκπαίδευση και εκπαιδευτικής πολιτικής. Έχουμε λοιπόν καταρτήσει αυτή τη σύνοψη της νομοθεσίας. Επικοινωνήσαμε και με εκπροσώπους του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών. Ανθρώπους λοιπόν στα κράτη-μέλη που ασχολούντουσαν με τα δικαιώματα των γυναικών. Ε, στο ε, έγγραφο αυτό το οποίο, το οποίο η πρώτη έκδοση εκδόθηκε το 2007 αλλά κατόπιν επικαιροποιήθηκε έχουμε εμείς ε, επισημάνει μία επιλογή έχουμε επιλέξει ποια είναι πλέον ε, ευνοϊκή για τις γυναίκες διάταξη και έκτοτε ε, συνεχίσαμε την προσπάθειά μας οργανώνοντας ένα συνέδριο υπό την Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 στην ε, στο οποίο παρευρέθηκε η Επίτροπος Μάλστρομ εκείνη την εποχή, υπεύθυνη για τα ζητήματα της ισότητας των δύο φύλων. Είχαμε επαφές με τα κράτη-μέλη, διμερείς, εκπροσωπήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ε, εκπρόσωποι των κρατών μελών παρευρήθηκαν στο συνεδρίο αυτό. συντάχθηκαν ε, προσχέδια συνθήκων, προσχέδια αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσπαθήσαμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα νομικά μέσα Καταγράψαμε επίσης θετικές και αρνητικές εξέλιξεις στα κράτη-μέλη σε σχέση με την ανάλυση του εθνικού δικαίου που είχαμε κάνει. Για παράδειγμα, ορισμένα. Έχουμε το παράδειγμα της Μάλτας, όπου το διαζύγιο δεν ήταν ε, ε, νόμιμο, δεν, δεν ήταν εφικτό, αλλά ε, αυτό ίσχυε τότε, το 2008, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, το διαζύγιο επιτρέπεται στη Μάλτα. Πιθανώς να υπάρξουν και άλλες εξελίξεις σε άλλα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, εξελίσσεται η συζήτηση για την έκτρωση. Προσπαθούμε λοιπόν να αναδείξουμε τα ε, θετικά σημεία στο θεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία ανέδειξαν το ζήτημα της ρήτρα της πλέον ευρωμημένης Ευρωπαίας. Ε, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέτρα του Στρασβούργου και περισσότερα κράτη-μέλη, υιοθέτησε το 2008 αυτή τη ρήτρα και δημιούργησε μια σχετική ομάδα εργασίας. Το Βέλγιο επίσης, η Βελγική ε, Γερουσία εξέτασε δύο προσχέδια απόφασης. στις οποίες θα αναφερθώ και πιο αναλυτικά αργότερα αν το επιθυμείτε και το Γαλλικό Κοινοβούλιο θέτησε σχεδόν ομόφωνα ένα ψήφισμα στις 22 Μαρτίου 2011 υπάρχουν και στη συνέχεια μάλλον αυτής της απόφασης στο Γαλλικό Κοινοβούλιο ζητήθηκε να μας δοθεί η δυνατότητα να επικαιροποιήσουμε την ανάλυση που είχαμε κάνει και αυτό τελικά οδηγεί και φτάνουμε στην συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που για μας είναι ιδιαίτερα σημαντική. όπως αναφέρατε και εσείς κύριε Αντιπρόεδρε, η κρίση στην οποία πλήττει τις χώρες της Ευρώπης, πλήττει επίσης και τις αξίες της και ιδανικά. Άρα θα επιθυμούσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μια συνέχεια μετά από τη σημερινή δημόσια εκρόαση στο έργο αυτό της ανταλλαγής ε, στοιχείων, κάτι που θα βοηθήσει και τους Ευρωπαίους πολίτες να έχουν μια αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται και με τα δικά του ζητήματα. Το 50% των πολιτών είναι γυναίκες, επομένως. Διαπιστώνουμε ότι και οι άνδρες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προσπάθειά μας και έχει τεθεί και το ζήτημα να γίνει κάτι αντίστοιχο για εκείνους. Λοιπόν, διαπιστώνουμε μια σύγκληση συμφερόντων και ενδιαφέροντος και το θεωρούμε σημαντικό. Όπως είπε και ο πρόεδρος Γκούσταυσον, έχει σημασία η ανταλλαγή των πρακτικών. Για παράδειγμα, Εάν δούμε πιο συγκεκριμένα τις διατάξεις για την αντιμετώπιση των περιστατικών βίας κατά των γυναικών, διαπιστώνουμε ότι το καλύτερο μοντέλο είναι εκείνο της Ισπανίας. Σε επίπεδο, η ανάλυση έχει γίνει σε επίπεδο Ευρώπης. Μια παρόμοια ανάλυση μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα ζητήματα. Θα επιθυμούσαμε να είναι ολιστική, όσο περισσότερο γίνεται. Γνωρίζουμε ότι τίθενται ζητήματα αρμοδιοτήτων και προβλήματα σχετικά. Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο της Νοντέρ διεξήγε μια έρευνα και θα μιλήσει πιο αναλυτικά για αυτό ο κύριος Σογό, ο καθηγητής Σογό, που θίγει ζητήματα που έχουν ασχολήσει την τελευταία δεκαετία υπουργικά συμβούλια, τους, ε, όλους εκείνους που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ίσως κάποια από τα ζητήματα λοιπόν εμπίπτουν πλήρως στις αρμοδιότητες τις νομοθετικές των κρατών μελών και άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Η κυρία έχει διεξάγει αυτή την έρευνα, καθώς επίσης και από τον οργανισμό μας η κυρία Ιμπού, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Το πρόγραμμα Ευκλήδης έχει δημιουργήσει το Πανεπιστήμιο της Νοντέρ με στόχο να συνεργάζονται φοιτητές και έτσι ώστε να υπάρχει μια μελέτη της, του προβλήματος σε συνεργασία με οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό. Σε Ίσως μίλησα πολύ για τη Γαλλία, αλλά το, πρόγραμμα είναι πραγματικά ευρωπαϊκό. Η Ιταλική αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας έχει βοηθήσει εξαιρετικά, στην, για παράδειγμα, στην μετάφραση και στην δημοσιοποίηση μέρων του ε, ανάλυσης του βιβλίου που εκδώσαμε στα Ιταλικά, στα Ολλανδικά. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω Έχει ξεκινήσει επίσης μια διαδικασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Συνθήκης, μιας Ευρωπαϊκής Έκκλησης, που φυσικά είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει. Έχουμε συνεργασία με πανεπιστήμια, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές συνέργειες, πολλές και σημαντικές συνεργασίες στην υλοποίηση του προγράμματός μας και τα διάφορα ε, στάδια του. Τι θα ε, αναμέναμε από εσά, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εκπρόσωποι του, των λαών της Ευρώπης, θα μπορούσε με, να ασκήσει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα πρωτοβουλία του και ευχαρίστω θα συνεργαστούμε μαζί σα εάν το πράξει αυτό. ακολουθώντας το παράδειγμα του, Συμβουλίου της Ευρώπης και του Γαλλικού Κοινοβουλίου να συνεργαστούμε με το Ινστιτούτο Βίνιους για να επικυροποιήσουμε την ανάλυση της αρχής νομοθεσίας που είχαμε κάνει. Μας φαίνεται εφικτό παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έλεγα μετά τις τρεις ε, παρεμβάσεις των ε, εμπειρογνωμόνων μας να ακούσουμε τις ερωτήσεις των βουλευτών και να έχουμε μετά τις απαντήσεις τους. Τώρα ο καθηγητής ε, Σωρών, κυβερνητικός σύμβουλος. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον κύριο Γκούσταυσαν για την πρόσκληση εδώ και να πω ότι είναι αλήθεια ότι θα προσπαθήσω με μεγάλη χαρά να εκφραστώ σε αυτήν εδώ την αίθουσα πριν από μερικά χρόνια όταν μου ζητήθηκε να ενταχθώ σε αυτή τη διαδικασία, θεώρησα ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και έβλεπα τις θετικέ πτυχές αυτής της ε, λεγόμενης ρήτας της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας. Το πραγματικό πρόβλημα σήμερα είναι, ότι η Ευρώπη ε, ε, ταυτίζεται για πολλούς ε, από τους πολίτες μας στην Ευρώπη με κάτι το αρνητικό. Μια πορεία προς τα πίσω. Αυτό είναι που παρατηρεί κανείς. Και πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο, η διαπίστωση ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πρέπει κανείς να παλέψει για όλα τα δικαιώματα για να μπορέσει να υπάρξει μια σύγκληση στις δράσεις. Τρεις μεγάλοι κατευθυντήρες γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν για αυτήν τη ρήτρα, για την πλέον ευνοημένη Ευρωπαία. Πρώτον, η χρήση ναι, όλων των ε, μέσων που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχει μια δυναμική. Το μείζον ε, θέμα, αυτά που είπε ο έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά απ' την άλλη υπάρχει αντίδραση ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει το α ή το β. Αντιστάσεις. Ε, πολλές φορές δηλαδή όλα χρησιμοποιούνται σαν πρόφαση να μην καταλήξει κάνει σε κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, οι συστάσεις τη επιτροπή, οι ε, συστάσεις του Συμβουλίου, δημιουργούν ένα τεκόρ ε, και βλέπουμε ότι δημιουργείται ε, ε, η αίσθηση ότι ξεκινάει κάτι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σιγά σιγά αναπτύσσεται. Αυτό μπορούμε να το έχουμε σαν δεδομένο. Φυσικά υπάρχει το θέμα που έχει να κάνει με τη νομική πτυχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά. Ε, έχουμε τη λεγόμενη μέθοδο ανοιχτού συντονισμού, όπου υπάρχουν ε, τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση όπου δεν έχει αρμοδιότητες, αλλά η πρόκληση δραστηριοτήτων σε, με ένα συντονισμένο τρόπο από τις χώρες μέλη. Και με αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια σύγκληση. Και επίσης κάτι το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία, η προσφυγή στην ενισχυμένη συνεργασία. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε να κάνουμε φυσικά αυτά σε κοινωτικό επίπεδο. Μετά έχουμε και το ε, εθνικό δίκαιο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει να κάνει με το, το θέματα που αφορούν συνθήκες όπου πολλές χώρες της Ευρώπης εντάσσονται. Ε, υπάρχει το λεγόμενο, η συνθήκη για τη λεγόμενη Σέγγεν 2, η οποία, συνθήκη η οποία, την οποία διαπραγματευτήκαν δύο χώρες, σε συνέχεια υπεγράφει από επτά και ένα χρόνο αργότερα εγκρίθηκε από τις 27 με τα πλαίσια μιας απόφασης πλαίσιο. Βλέπουμε δηλαδή πόση σημασία έχει όταν, ε, πόση μεγάλη σημασία έχουν διμερείς φερρυπίν αποφάσεις και πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικότατο στις, ε, ε, στο αυτό που έχει δημιουργηθεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας μέσα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Το 2014 αφερπίν. οι μεγάλες πολιτικές ομάδες θα ορίσουν, κάνουν ένα διορισμό και, και στα πλαίσια αυτά είναι εμείς που πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια ε, για να οδηγηθούμε ε, σε μια Ευρωπαϊκή Προεδρία, όπου εδώ μπορούμε να δούμε μια ρήτρα η οποία να είναι ανάλογη με το θέμα που μας αφορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε ένα διάλογο, ε, πολιτικό διάλογο, στα πλαίσια της επόμενης Επιτροπής και ελπίζουμε αυτός ο διάλογος να είναι όσο δυνατόν πιο ανοιχτός. Δεύτερο στοιχείο. Η, πρωτα, η πρωτοβουλία για την ε, ευρωπαϊκή υπηκότητα. Ξέρουμε ότι χρειάζεται η πρωτοβουλία αυτή χρειάζεται την υποστήριξη ενό εκατομμυρίων υπογραφών. Φαίνεται ότι είναι σημαντικό, αλλά σε επίπεδο συνδικαλιστικό, φερρυπίν σε κινητοποίησεις είναι εφικτό. Ε, Έχουν να κάνουμε εδώ με προβληματισμούς οι οποίοι δεν περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά πιάνουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά είναι σημαντικά. Να δούμε δηλαδή την Ευρώπη σαν κάτι περισσότερο από σύνολο εθνικών δικαίων. Επίσης, κάτι που είναι τεχνικής ίσως φύσεως, έχουμε να κάνουμε μια ρήτρα επιτάχυνσης που επιτρέπει σε ορισμένους τομείς ε, αυτά τα οποία είναι τα πιο δυναμικά θα λέγαμε κράτη να επιταχύνουν τις διαδικασίες, να εγκρίνουν ένα κείμενο αφότου διαπιστώσουν ότι μπορεί να υπάρξει συνέχεια η δυνατότητα να εγκριθεί από τις 27. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι δεν υπάρχει ένα μόνο δίκαιο, όχι ένα μόνο μέσο. Θα πρέπει να προβληματιστούμε σε επίπεδα στρατηγικής, στρατηγική πώς θα βρούμε μέσα και επίπεδα δράσης και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε μόνο, μόνο, μόνο κεντρικά στην Ευρώπη θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ε, εθνικό επίπεδο, διότι και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε πρόοδο. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον Ζαλίξορο. Πολύ καλή παρέμβαση, συγκεκριμένη. Μας αναφέρει τις ε, νομική ε, διάστασης προοπτικές. Θα, δώσω το λόγο στη κυρία Βελό. Thank you very much for the uh, σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Έχω να σας κάνω μια παρουσίαση σε PowerPoint. Είναι τιμή μου που είμαι προσκεκλημένη εδώ και πρέπει να πω ότι εγώ ίδια ωφελήθηκα, δεν είχα ακούσει ποτέ για τη ρήτρα αυτή να προσκληθώ σε αυτή την ακρόαση και είμαι εξειδικευμένη στα θέματα ισότητας των δύο φύλων. Φαίνεται Λοιπόν, από ερευνήτρες όπως εγώ, ότι αυτό το θέμα έχει αποκρυπτεί, ε, χαίρομαι πολύ που το έμαθα λοιπόν. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα καινοτόμο εργαλείο. Ένα εργαλείο που έχει οδηγήσει στην ε, δημιουργία διαλόγου σε εθνικό, τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλαπλασιάζονται λοιπόν οι προσπάθειες που θα έπρεπε να κάνουν και κάνουν ε, όλοι για την ισότητα των φύλων. Στον ε, τίτλο μου χρησιμοποιώ τον τίτλο ε, «Ισότητα των φίλων περισσότερων του ενός» διότι η ισότητα των φύλων δεν πάει ποτέ μόνη της. Μπορεί να έχει να κάνει με την σεξουαλική ανισότητα, με την ε, ανισότητα σε, άλλα, σε άλλους τομείς. Εδώ λοιπόν αναζητούμε θεσμικούς μηχανισμούς και πού αυτή η ρήτρα θα μπορούσε να ενταχθεί. για τις αρχές της ανισότητας. Έχουμε εντοπίσει κάποια θέματα στις διαδικασίες. Εάν θέλουμε μηχανισμοί να είναι αποτελεσματικοί, θα πρέπει να δίνουμε περισσότερη, περισσότερες σημαντικότητες, περισσότερη εξουσία στους ε, υπέρμαχους της ισότητας των γυναικών. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί και οι μηχανισμοί. Επίσης για τις διαδικασίες. Υπάρχει άμεση ανάγκη για δράση, αλλά και για διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα να επιτευχθεί πρόοδος σε σχέση με το ποιο είναι το σκηνικό που επικρατεί σε κάθε διαφορετική χώρα. Όταν μιλάμε λοιπόν για νομικούς και θεσμικούς μηχανισμούς θα πρέπει το σκέλος της ισότητας των φύλων να είναι κάτι που προβάλλεται, που είναι ορατό. Πολύ λόγου χάρη είναι οι σύλλογοι που ζητούν την προστασία των εργαζομένων σε μερική απασχόληση. Συνήθως είναι γυναίκες αυτές, αλλά θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στο gender plus να διατηρηθεί αυτό το πρόσημο, το θετικό πρόσημο. Και εδώ <clears throat> να προσπαθήσουμε να μετατρέψουμε θετικά τις κοινωνίες μας, χάρη στη διάσταση αυτή. Εάν δούμε τους νομικούς και θεσμικούς μηχανισμούς, νομίζω ότι είναι τρία τα βασικά σημεία που μας ενδιαφέρουν. Πρώτα απ' όλα οι νόμοι και οι κανονισμοί. Ένα σύνολο κανόνων σε γενικές γραμμές. Είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά. Τα υπόλοιπα δύο είναι πρώτα απ' όλα οι ίδιοι οι άνθρωποι και το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή πώ διοργανώνονται ώστε να επιδιώξουν την ισότητα των φύλων. Εδώ μιλάμε για φορεί, φορεί που ασχολούνται με τι πολιτικέ που αφορούν τι γυναίκε, την ισότητα των φύλων, τι υπηρεσίε, του οργανισμού που λαμβάνουν αποφάσει που μπορεί να ε, είναι υπέρμαχοι και να υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Και ένα άλλο σκέλο είναι οι πόροι, τα κονδύλια, τα χρήματα, ο χρόνο, οι ευκαιρίε που υπάρχουν για να επιδιωχθούν η ισότητα των γυναικών. Επίσης, να τονίσω ότι πάντοτε υπάρχει μια ποικιλία στρατηγικών και θεσμικών ε, οργάνων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Είναι πολυδιάστατο το φαινόμενο. Την ισότητα την θετική ισότητα των φύλων μπορούμε να την πετύχουμε μόνο με συνδυασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Κάποιε είναι πιο αποτελεσματικέ προ μια κατεύθυνση και κάποιε προ μια άλλη. Πρέπει όμω και τι δύο κατευθύνσει να τι επιδιώκουμε ταυτόχρονα. Χρειαζόμαστε την δράση και θετικέ συστάσει για να πετύχουμε κάτι. Επίση, μπορεί κανεί να πετύχει αυτή την ε, θετική ισότητα των φύλων με το συνδυασμό ε, προληπτικών και μέτρων και μέτρων που προωθούν την δράση. Κάποιε φορέ οι γυναίκε υποφέρουν από τι ανισότητε και πρέπει να του προσφερθεί προστασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όμω πρέπει κανεί να λάβει και δράση προκειμένου να αλλάξει η κατάστασή του που τη θυματοποιεί. Δύο συνάδελφοί μου που εργάζονται για το θέμα αυτό τη ε, θετική ισότητα των φίλων λένε ότι το θέμα αυτό μοιάζει με την, ισότητα, με την Λερναία Ήδρα. Κόβει ένα κεφάλι και γεννιέται ένα άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε καλύτερε στρατηγικέ για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το θέμα. Επ' αυτού, είτε μιλάμε για του καλύτερου νομικού ή θεσμικού μηχανισμού, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα δύο πράγματα ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ότι πάντοτε θα πρέπει να είμαστε αρκετά τολμηροί ώστε να βλέπουμε τι είναι αυτό που θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο και να το δηλώνουμε ανοιχτό και να συνειδητοποιούμε ότι ίσως εάν αλλάξει το γενικότερο σκηνικό αυτό που είναι το καλύτερο μπορεί να μεταβληθεί. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει διαρκή συνεχιζόμενος διάλογος για τα θέματα αυτά. Νομίζω σε ό,τι αφορά τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς η ρήτρα της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας είναι μια θαυμάσια πρωτοβουλία. Και αυτό γιατί τονίζει τις καλύτερες, τις σημαντικότερες προτεραιότητες των όσων θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε. Πολλαπλασιάζει τα θετικά παραδείγματα και ουσιαστικά μας κάνει να αποφύγουμε την ε, επικίνδυνη προοπτική του ελάχιστου κοινού παρονομαστή. Στο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο ηγούμε τα τελευταία χρόνια, το πρόγραμμα που υπάρχουν πολλά παραδείγματα και σε τοπικό επίπεδο. Σκεφτείτε τι γίνεται στη χώρα των Βάσκων, την Καταλωνία, την Φλάνδρα, την Ουαλία, τη Σκοτία. Υπάρχουν ε, παραδείγματα και σε εθνικό επίπεδο άλλε φορέ. Εάν η Ισπανία αντιμετωπίζει τόσο καλά τη βία, αυτό οφείλεται και στο δυναμικό χαρακτήρα των διαφορετικών ε, επαρχιών και το πώ συνδυάζονται τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο για να φτάσουν στο εθνικό. Επίση, το θέμα δεν είναι μόνο πόσο καλή είναι οι νόμοι και οι κανονισμοί, αλλά αν και πραγματικά επιβάλλονται, αν ε, εφαρμόζονται. Πώς δηλαδή το κράτος μπορεί να ελέγχει εάν αυτά που προβλέπει ο νόμος ισχύουν και εφαρμόζονται τι γίνεται στην πραγματικότητα και πώς οι πολιτικές διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων μπορεί να αντικατοπτρίζονται σε αυτή τη ρήτρα. Νομίζω είδαμε παραδείγματα στην ε, Ολλανδία όπου για την πορνεία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις λόγου χάρη. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι μια θέση είναι καλύτερη από άλλη και πρέπει να επιδιωχθεί και να αναλυφθεί δράση. τώρα να έρθω σε μια πρόταση για το πώς θα μπορούσαν τα θετικά στοιχεία να εξερευνηθούν και να αξιοποιηθούν καλύτερα. Πώ μπορούμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Αν δούμε του ανθρώπου και το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχει ανάγκη να σκεφτούμε περισσότερο κατά πόσον οι φορεί που επιδιώκουν την ισότητα των γυναικών και οι φορείς που ασχολούνται με την θετική ισότητα των γυναικών είναι αποτελεσματικοί. Σε όλη την Ευρώπη βρίσκουμε ότι οι φορεί αυτοί αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα, είναι σε σύγχυση. Ε, στις, στην περίπτωση της Βρετανίας, λόγω χάρη, υπάρχει θέμα ανισότητας με τι γυναίκες. Κάποιες φορές ε, τα μέλη σε επιτροπές της Βουλής δεν ε, εκπροσωπούνται αρκετά από γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το σχήμα που λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Στο δικό μας το πρόγραμμα είδαμε ότι η ιδανικότερη μορφή ως τώρα δεν είναι να έχουμε ένα θεσμικό όργανο ενιαίο αλλά ένα όργανο όπου υπάρχουν διαφορετικοί πιλότες για να αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι ανισότητες και να υπάρχει ένας διαρκής διάλογος μεταξύ αυτών των πυλώνων. Παρομοίως, είδαμε ότι σε ό,τι αφορά τους θεσμικούς μηχανισμούς σε κάποιες χώρες δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πια συμβουλευτικοί φορείς για την θετική ισότητα των φύλων. Οι κάτω χώρες, συμπεριλαμβάνονται τις χώρες αυτές, υπήρχε Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων και σχετικό συμβούλιο, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη. Διότι οι προσπάθειες για τα γυναικεία δικαιώματα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να επιδιώκονται με την απουσία φορέων. Χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό που να συνοδεύει τους νόμους και κανονισμούς. Παρομοίως, αυτό ισχύει και για τους πόρους, που είναι ένα σημαντικό νομικό και θεσμικό εργαλείο. Κάποιοι έχουν κονδύλια για την ισότητα των φύλων και έχουν μια πολύ σαφή αντίληψη του πώς ε, αποδίδουν ε, τα κονδύλια αυτά στις προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας. Συνοψίζοντας, η ρήτρα, πιστεύω, είναι πολύτιμη πρωτοβουλία Πρέπει να προσπαθήσουμε να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της σε όλη την Ευρώπη, αλλά και να επεκταθεί η χρήση της. Κάποια στοιχεία αυτή τη στιγμή που αφορούν τα κονδύλια, τους πόρους, όπως για την άμβλωση, είναι σημαντικά και στην Ολλανδία έχουμε ένα σχετικό παράδειγμα. Για ορισμένους προβλέπεται δωρεάν πρόσβαση. Επίσης, σωστά παρακολουθούνται οι νόμοι και οι κανονισμοί, οι φορείς και συγκεκριμένα παραδείγματα. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσε αυτό να γίνει συνολικότερο και να επεκταθεί. Merci euh, à vous. Merci de... Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας δώσετε τη δική σας προσέγγιση στα πράγματα. Και έτσι συνοπτικά. Αξιοποιήσατε κατά το χρόνο που σας δόθηκε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επανέλθω προσπαθώντας να θέσω και το πλαίσιο της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Στο εξή, αυτό που μας απασχολεί εδώ, στη βάση του, είναι η ισότητα των πολιτών της Ένωσης. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η ρήτρα της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας είναι μια μάχη φεμινιστριών με άλλους. Εμείς το ανταλαμβανόμαστε ως ένα μέσο για να εξασφαλίσουμε την ισότητα όλων των πολιτών στην Ευρώπη. Και έτσι πρέπει να ε, εξετάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα. Θεωρώ ότι το έργο της Επιτροπής εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Επιτροπής μας, ε, επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτήν την λογική της προάσπισης της ισότητας των πολιτών. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω είναι ότι υπό τη ρήτρα της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας μπαίνουν πολλά θέματα και πολλά από αυτά απασχολούν ιδιαίτερα την Επιτροπή μας. Σίγουρα θα αναφερθούν και συνάδελφοι. Για παράδειγμα αναφέρομαι στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που αποτελεί και παραβίαση στην αρχή της ισότητας, οι ανισότητες στην αμοιβή, στη, για την εισεργασία. Σας δίνω μόνο δύο παραδείγματα στα οποία η Επιτροπή μας έχει ιδιαίτερα επισταμένα ασχοληθεί. Επίσης έχουμε συνεργαστεί, αν και μένουν πολλά ακόμα να γίνουν, προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή την συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση, όχι μόνο δηλαδή μια προσέγγιση νομική, αλλά επίσης και συνολικά στατιστικά στοιχεία που θα μας δίνουν μια ακριβή εικόνα, μια φωτογραφία των ανισοτήτων που υφίστανται που ε, στο ένα ή στο άλλο τομέα μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, σήμερα βλέπουμε το... και εξετάζουμε τον αντίκτυπο της κρίσης την εργασία των γυναικών και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια έλλειψη στατιστικών στοιχείων, ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τις τελευταίες εξέλιξεις. Άρα, με χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας στο σύνολο αυτών των ζητημάτων ο λόγος τώρα στα μέλη της Επιτροπής. Βλέπω ότι η Μαρία Καπριέλ ε, έχει ζητήσει το λόγο. Τον, σας τον δίνω παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστώ που οργανίσατε αυτή την ακρόαση η οποία πραγματικά μπαίνει στην καρδιά του θέματος, θεμάτων που αφορούν ε, τη δική μας Επιτροπή και ε, φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θεωρώ ότι η ρήτρα για την οποία συζητούμε μας κάνει να καταλάβουμε και κάτι το οποίο υπεγραμμίσει από τους προλαλήσαντες ε, μας οδηγεί σε διαπίστωση ότι υπάρχουν και πρόοδοι αλλά και υποχωρήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών. Φυσικά υπάρχει το θέμα των βέλτιστων πρακτικών και το θέμα της αξιολόγησης αυτών των πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και κοινωτικό επίπεδο. Θα, μείνω πιστή πιο πολύ σε αυτά τα οποία ε, ήταν προσφυλή πριν να μπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά να πω ότι υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία. Το ένα έχει να κάνει με τον βαρικό χαρακτήρα της ρήτρα. Όταν μιλάμε για την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ρήτρα είναι ότι μιλάμε για διαφορετικές πρακτικές σε χώρες μέλη που τείνουν να ενισχύσουν τη θέση της γυναίκας σε κάθε χώρα. Το πρόβλημα για μένα είναι το εξή. Πρώτον, η, επι... η επιλογή ενός μοντέλου και δεύτερον, την διάδοση αυτού του μοντέλου. Καταρχήν λοιπόν έχουμε να κάνουμε τη μελέτη των διαφορετικών μοντέλων, να δούμε τις επιπτώσεις τους, να δούμε πώς συμβάλλουν σε θέματα των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά κυρίως να επιλέξουμε το καλύτερο από αυτά, ούτως ώστε να το εγκρίνουμε, υιοθετήσουμε και να διαδώσουμε. Αυτή η μέθοδος μου φαίνεται ότι είναι η καλύτερη μάλλον για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια αποτυχία. Οι, οι πρωτοβουλίες είναι πολλές και ακούω συχνά ότι τα θέματα των, ε, που είναι γυναικείου ενδιαφέροντος δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσει κανείς ε, με ένα και μόνο τρόπο. Κάθε γυναίκα έχει τη δική της πραγματικότητα και γι' αυτό το λόγο η, η ρήτρα για την οποία συζητούμε πρέπει να δώσει έμφαση σε κάποια σημεία τα οποία θίξαν οι προλαλήσαντες και μας δίνουν μια κοινή εκκίνηση για να καταλήξουν σε κάτι πιο συγκεκριμένο και κοινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτον, να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τις πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τις ισότητες των φύλων. Στη συνέχεια να δούμε τα, τις ανάγκες των γυναικών σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο. Στη συνέχεια να εντοπίσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που τις εμποδίζουν να μπορέσουν να ανασκήσουν τα δικαιώματά τους και δεύτερον η δημιουργία ενός δικτύου βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Καθηγήτρια, επιμείνατε πολύ στο θέμα του συντονισμού που είναι απαραίτητη τόσο σε εθνικό όσο και κοινωτικό επίπεδο. Το Ινστιτούτο το Ευρωπαϊκό για τα, την ισότητα των φύλων μας είναι σημαντικό γιατί κάνουμε συγκεκριμένα κάποια πρόοδο πάνω σε αυτό και βάσει σε αυτές τις τέσσερις πτυχές μπορούμε να πετύχουμε ίσως ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και κυρίως ότι θέτει σε έμφαση την προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Δηλαδή, η ενότητα μέσα στην πολυμορφία. Αυτό θα πρέπει να το βλέπουμε. Κάτι ακόμα το οποίο όπως ε, ελέγχθη είναι ε, αυτό που έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες και φυσικά τα μέσα, τα κονδύλια για την ε, εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε στην Επιτροπή τη δική Το πρώτο που με ενδιαφέρει είναι ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας της ρήτρα αυτή Μοντέλο, διάδοσή του, δεύτερον στρατηγική. Αυτή η ακρόαση οργανώθηκε ακριβώς για να εντοπίσουμε βήματα σταθερά που μπορούν να μα οδηγούν σε πρόοδο. Όπως είπε η κυρία καθηγήτρια, μα είπε ότι ο δρόμος είναι μακρύς, ε, είχαμε όλη την προσπάθεια που κατέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα και σήμερα το θέμα τίθεται ως εξής. Πώς μπορούμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτή την ιδέα της ρήτρα, κάτι απτό. Εντυπωσιώστηκα από τις προτάσεις του συγκεκριμένου του κυρίου Σωρών η ιδέα που έχει να κάνει με τον υποψήφιο για την Προεδρία της Επιτροπής της επόμενης. Καλό είναι να εκφραστεί πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τη πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών είμαι λίγο επιφυλακτική. Έχει γίνει κάτι τέτοιο και έχει γίνει πρωτοβουλία από νέους, αλλά βλέπουμε στην πράξη πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει κανείς. Γι' αυτό αναρωτιέμαι αυτό το θέμα της συμμετοχικής δημοκρατίας πώς μπορεί να οδηγήσει στο να προσθέσουμε. Στα πλαίσια της συνθήκης της Αβώνας πάντα, έχω κάποιες επιφυλάξεις. Ε, έχω επιφυλάξει παρόλο που εγώ είμαι πολύ ενθουσιασ... Ε, από τους θετικούς όσον αφορά αυτές τις πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι πώς θα μπορούσε αυτό να είναι μέσω στα χέρια του Ευρωπαίου πολίτη τους ώστε να κινητοποιηθεί και να προβληματιστεί να βρει νέα μέτρα μέσα. Θα ήθελα να πω επίσης και αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε στην διάδοση ε, όταν γίνονται κάποιες δράσεις. Υπενθυμίζω ότι διάφορες χώρες οι οποίες έχουν ε, δραστηριοποιήσει το θέμα της, ε, του διαζύγιου Φερρυπίν και θέλουν να προχωρήσουν πιο πολύ από τις άλλες. Αλλά αυτό το θέμα δεν είχε μεγάλη απήχηση. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουμε εκτός από τα μέσα που αναφέρατε και προτείνατε. Και θα ήταν καλό να δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας από Ευρωπαίους ε, Ευρωβουλευτές και σε συνεργασία με εθνικούς βουλευτές να προβληματιστούν πραγματικά και να δούνε τις σημαντικές πτυχές των θεμάτων που είδαμε εδώ σήμερα, ούτω ώστε αυτή η ρήτρα να κατά κάποιο τρόπο να φύγει από το πλαίσιο αυτό το καθαρά θεωρητικό και να δούμε ούτως ώστε να γίνει μια πρωτοβουλία η οποία πρέπει να οδηγηθεί σε ε, ε, κοινοτικό επίπεδο. Άρα, ομάδα εργασίας η οποία θα μας επιτρέψει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα στα πλαίσια των επόμενων ευρωεκλογών. Ευχαριστώ. Merci à Maria Gabriel. Ευχαριστούμε τη Μαρία Γκαμπριέλ για την ανάλυση της και την θεώρησή της για το πώς μπορεί να μεταβληθεί η ιδέα σε πράξη. Η Edith Bauer και μετά η Bill Thompson. Ίσως η Edith Bauer πρώτη και μετά η κυρία Thompson. Edith. Madame Thompson. Alors, Madame Thompson, pas de problème. Thank you very much. Κυρία Τόμσεν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία να διοργανωθεί αυτή η ακρόαση που είναι σοβαρότατη. Πραγματικά την πρώτη φορά που άκουσα για, την, για το βιβλίο αυτό της ε, κυρίας της ε, Κυρία Διπανή για τη ρήτρα τη πλέον ευνοημένη Ευρωπαία, εντυπωσιάστηκα πραγματικά για τα θέματα ισότητα των φίλων που συζητάμε εδώ στην Ευρώπη. Προφανώ ενδιαφερόμαστε όλοι, αλλά είναι ένα πρότυπο που θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε σε όλου του τομεί. Θα μπορούσαμε να είμαστε εμεί οι πρωτοπόρε και να έχουμε επινοήσει εμεί το μοντέλο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχουμε παράδοση στα θέματα των φύλων. Ανέκαθεν είμαστε μπροστά από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν ισχύει για όλους τους πολιτικούς τομείς, διότι συνήθως οι πολιτικοί ηθήνοντες δεν βρίσκονται στην εμπροστοφυλακή. Πρώτα λαμβάνουν χώρα εξελίξεις και μετά το συνειδητοποιούν οι πολιτικοί. Σε ό,τι αφορά όμως την ισότητα των φύλων, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουμε ξεπεράσει τα κράτη-μέλη. Βεβαίως, το 2006 μας ξεπέρασε η Ισπανία που υιοθέτησε σχετική νομοθεσία. Όμως να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση της εμπροστοφυλακής, εμπνέοντας τα κράτη-μέλη. Νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό εν ώψη της στρατηγικής του 2020 για την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη και τα θέματα των φύλων διότι ζητούμε το 75% των εργαζομένων στην εργασία αγοράς να παραμένουν ενεργοί αν θέλουμε να διατηρήσουμε το κράτος πρόνοια στην Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι 76% των ανδρών είναι ενεργοί στην ε, αγορά εργασίας. Το πρόβλημα τίθεται με τις γυναίκες. Μόνο το 60% περίπου είναι ενεργές. Θα πρέπει εδώ να ανταλλάξουμε εμπειρίε και ιδέε για το πώ μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στην ε, αγορά εργασία οι γυναίκε, αλλά και την, ε, ε, με την ανατροφή των παιδιών πρέπει να ασχοληθούμε, με την μέρημνα για τα παιδιά. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τι γυναίκε και να εργάζονται και να φροντίζουν την οικογένειά του. Είναι μια βασική ανάγκη αυτή για όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι να απευθυνθούμε στο Ίδρυμα για την Ισότητα, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των ε, φίλων είναι μια καλή ιδέα. Θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε σταδιακές για τις διαφορετικές χώρες και πιστεύω για άλλη μια φορά ότι από κοινού μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Είναι κάποιοι τομείς όπου σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τα ίδια θέματα. Όπως το θέμα της ε, πορνείας που αναφέρετε κι εσείς για την Ολλανδία. Στις σκανδιναβικές χώρες το θεωρούμε κάτι το απέσιο, υποβαθμιστικό για τις γυναίκες. Αυτή είναι η δική μας η αντίληψη. Αλλά σε άλλες χώρες όπως η Δανία, βασικό πρόβλημα της ισότητας των φύλων είναι το να αναγνωριστούν και οι βασικές διαφορές μεταξύ των φύλων. Στην στην ε, Δανία που πήγα τελευταία έτυχε να με σερβίρει ένας ε, άντρας και είπα ότι σπάνια συμβαίνει αυτό σε έναν ε, τέτοιο χώρο και εκείνος μου απάντησε «Μα κοιτάξτε, δεν είμαστε στη Δανία, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα». Να κάτι που θα μπορούσε να συμβαίνει και άλλο στην Ευρώπη. Επίση, για τα κράτη-μέλη, νομίζω η μέθοδο ανοιχτού συντονισμού είναι μια καλή ιδέα. Η μέθοδο που ανέφερε ο κ. Σωρών. Ανυπομονώ λοιπόν να συνεχίσουμε τη δουλειά μα για τη ρήτρα τη πλέον ευνοημένη Ευρωπαία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμψεν για τις δικές σας σκέψεις και ανάλυσεις και επίσης για την προσήλωση που έχετε επιδείξει στο ζήτημα. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που διοργανώσετε αυτή τη δημοσιοκρόαση και την ανταλλαγή απόψεων. Ξεκινώ λέγοντας απολύτως ειλικρινά ότι είμαι ελαφρώς προβληματισμένη, μπερδεμένη από αυτή την ε, έκφραση ρήτρα της πλέον ευνοημένης, πλέον ευνοημένης ε, Ευρωπαίας. Δεν θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να διοργανώσουμε κάποιου τους διαγωνισμό σε, τόσους τομεί, σε, σε διαφορετικούς τομείς, γιατί η νομοθεσία καλύπτει πολλούς διαφορετικούς τομείς και είναι δύσκολο κανείς να συγκρίνει για παράδειγμα τον τομέα της βίας που εμπίπτει στο ποινικό δίκαιο ή άλλα τομείς που οποιου στους οποίους αναφερθήκατε, οι οποίους εμπίπτουν στο εργατικό δίκαιο ή άλλοι που εμπίπτουν στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η μητρική άδεια ή άδεια λοχίας. Βλέπετε αδεια είναι ξεχωριστή τομείς και ίσως εγώ να μην αντιλαμβάνομαι σωστά Ποια ήταν η ιδέα, ποια είναι η λογική. Αλλά αφού θέτουμε το ζήτημα από πλευράς φίλου ή gender plus φίλου και πλέον, θεωρώ ότι μπορούμε να το, να το εξετάσουμε σε εξής. Υπάρχει ένα πολύ καλό νομικό θεσμικό πλαίσιο το οποίο όμως δεν είναι επαρκές. Όταν για παράδειγμα τίθεται το ζήτημα της νομικής αποζημίωσης. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις στα διάφορα κράτη-μέλη. Σε ορισμένες ε, περιπτώσεις, για παράδειγμα, η νομική βοήθεια παρέχεται δωρεάν. Σε άλλα κράτη-μέλη, μπορεί τα θύματα, να, οι γυναίκες να έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ υψηλό κόστος για να ασκήσουν ένδικα μέσα και να δυσκολεύονται να προσφύγουν στο νομικό, στο δικαστικό σύστημα. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε για τα σφορείς, για την ισότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε στη διάθεσή σας κάποιες αναλύσεις, στοιχεία σε αυτόν τον τομέα. Γιατί σύμφωνα με την νομοθεσία, κάθε κράτος μέλος πρέπει να έχει ένα φορέα για την ισότητα. Αλλά πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η φορείς, ποιες αρμοδιότητες έχουν. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε μια ανάλυση να δούμε τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Μήπως δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για την αντιμετώπιση της, του προβλήματος. Υπάρχουν άλλα. Άλλα εργαλεία. Αναφέρθηκαν ορισμένα, όπως για παράδειγμα η ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών η μέθοδος ανοιχτού συντονισμού. Αλλά όχι, όχι σε αυτό τον τομέα. Όχι, ακόμα τουλάχιστον. Σε ορισμένες περιπτώσεις η νομοθεσία των κρατών είναι πολύ διαφορετική. Το διαπιστώσαμε, για παράδειγμα, στο ζήτημα της μητρικής άδειας. Είναι τόσο διαφορετική η νομοθεσία στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μάλλον δεν θα καταφέρουμε ούτε καν να εξυγχρονίσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία γιατί βασίζεται σε κοινωνικά μοντέλα και συστήματα χρηματοδότησης πολύ διαφορετικά. Είναι δύσκολο ακόμα να, να, να βρεθεί ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής ακόμα και σε αυτό το τομέα μεγάλο αυτό το ζήτημα, δεν θέλω να το ανοίξω στο, σύνολό του. Απλώς συνοψίζοντας, θέλω να ρωτήσω τι έχετε διαπιστώσει εσείς στον τομέα πρώτον των ενδίκων μέσων και δεύτερον των φορέων για την ισότητα. Και ζητώ συγγνώμη για τη, μη παρουσία μελών της Επιτροπής. Πολλά ε, μέλη ήταν ε, υποχρεωμένα να πάνε σε άλλες επιτροπές γιατί υπήρχαν ψηφοφορίες. Ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Πριν δώσουμε και πάλι το λόγο στις εμπειρογνωμόνες και στους εμπειρογνωμόνες, να δώσω την ευκαιρία στην Πέτρα Σότ να παρέμβει, πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας και για την παρουσία σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο. Εργάζομαι στον τομέα της νομικής υπηρεσίας και δικαιοσύνης για τα θέματα ισότητας των φύλων. Έχουμε συμμετάσχει στην επεξεργασία των ε, μεζώνων οδηγιών τα τελευταία χρόνια για την οδηγία λόγω χάρη για την ε, ποσοστώσει, την οδηγία για τις άδειες μητρότητας που αναφέρθηκε εδώ, τη γονική άδεια, την ε, άδεια μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες, παραδείγματα την περσινή μόνο χρονιά. Επίσης, είμαστε σε επαφή με τον δικό σας οργανισμό, την ε, ρήτρα της πλέον ευνοημένης Ευρωπαίας, θεωρούμε ότι είναι πολύτιμο το έργο σας γιατί αφορά τις βελτιστές πρακτικές. Αυτό κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν σχεδιάζει νέες νομοθετικές προτάσεις. Κοιτάζουμε τι ισχύει στην Ευρώπη και τι θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φυσικά οι απόψεις πολλές φορές είναι διαφορετικέ και αντικρώμενε. Δεν μπορούμε πάντοτε να επιλέξουμε την ιδανική λύση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ε, έχουμε αρμοδιότητα από τις ε, συνθήκες να επιδιώκουμε την ελάχιστη εναρμόνιση. Δεν μπορούμε πάντοτε να επιζητούμε τα πλέον δαπανηρά, τις πλέον δαπανηρές λύσεις. Πρέπει να σεβόμαστε και τα όρια που μας ε, θέτουν οι συνθήκες. Μια σχετική εναρμόνιση λοιπόν Και εκεί ακριβώ κάπω αποκλίνουν οι απόψεις μας, διότι εμείς υποχρεούμαστε να τοποθετηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο, ενώ ένας ερευνητής αναζητά την ιδανική λύση, την βέλτιστη νομοθετική λύση ή διαδικασία για τις γυναίκες. Πάντως το έργο σας είναι πολύτιμο και για μας, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι έχουμε μια ποικιλία απόψεων. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το θέμα, αλήθεια είναι αυτό όπως είπατε. Να εντοπίσουμε τέτοιες καλές προσπάθειες, διότι οι δημοσιονομικές νοοτροπίες, οι νομοθετικές νοοτροπίες στα κάτι μελη διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Η καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ας πάρουμε το παράδειγμα της άδεια μητρότητας λόγου χάρη. Ή το τι γίνεται με τις διατροφές μετά από ένα διαζύγιο. Ή την ε, ε, γονική μέρημνα, την τη διεκδίκηση ενός παιδιού μου από το ένα διαζύγιο. Κοιτάζουμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει με την περίπτωση της ρήτρα και αν είναι καλύτερα να, έχουμε, να επιδιώκουμε την ιδανική λύση ή μια λόγω χάρη μικρότερη περίοδο αλλά με καλή αμοιβή. Είναι σημαντικό πάντως όπως είπατε και εσείς να έχουμε μια εικόνα συνολική. Κάτι σαν πανόραμα. Αυτό προφανώς είναι πολύτιμο και για μας. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε. Να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στι εμπειρογνώμονε, αλλά με αντίστροφη σειρά από τη σειρά που σα ακούσαμε. Η κυρία Βερλό. Θεωρώ πολύ χρήσιμα αυτά τα σχόλιά σας γιατί θα ξεκινήσω και από τις τελευταίες ε, παρεμβάσεις ε, ίσως αφηρημένα να είναι πολύ καλό και εύκολο να μιλάει κανείς για τον, την βέλτιστη πρακτική, αλλά χειροπιαστά και συγκεκριμένα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό, αυτό λέτε. Αυτό που πρέπει να μην ξεχνούμε είναι ότι πάντα υπάρχουν δύο διαφορετικές επιλογές. Η πρώτη είναι η πολιτική διεκδίκηση. Εδώ πρόκειται για έναν φορέα δημοκρατικό που λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία, επομένως μπορεί κάποιο να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του, να αγωνιστεί να επιδιώξει το καλύτερο για ε, εκείνον. Η δεύτερη επιλογή είναι εκείνη που βασίζεται στις αξίες. Εκεί, κάνοντα για παράδειγμα μία ε, μελέτη των ε, διατάξεων για τη γονική άδεια σε ολόκληρα τα κράτη-μέλη μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι καμία από αυτές τις διατάξεις, από αυτές τις νομοθεσίες δεν είναι επαρκώς, δεν, η επαρκής, δεν είναι η καλύτερη, με βάση τις αρχές τις οποίες βασίζεται. Ε, άρα θέτει κανείς συγκεκριμένα κριτήρια για την έρευνά του, με διαφάνεια, και διεξάγει έτσι αυτή την έρευνα ή επιλέγει την οδό της ε, λήψεις αποφάσεων μέσω των δημοκρατικών οργάνων. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύτιμο να αξιοποιηθεί η ρήτρα όσο έχει σήμερα. Μπορεί φυσικά να τροποποιηθεί στο μέλλον, αλλά έχει νόημα κατά την άποψή μου να ξεκινήσει αξιοποιώντας αυτή τη ρήτρα μια συζήτηση, μια δημόσια συζήτηση για να εξευρεθεί ποια είναι η βέλτιστη πρακτική. Και αυτό από μόνο του κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα ε, αποτελεσματικό. Δεν θεωρώ ότι το να συζητούμε και να αναζητούμε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή θα μας οδηγήσει πουθενά. Αυτό δεν έχει αξία. Αυτό που έχει αξία είναι να πολλαπλασιάσουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες ε, πολιτικών, πολιτών, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες λύσεις. Και αυτό θα γίνει μέσα από φόρουμ διαλόγου. Σε αυτό εγώ θα ε, εστίαζα. Πολλοί αναφέρθηκαν στο Ινστιτούτο ε, Ισότητας των Δύο Φίλων στο Βίλνιου και το ρόλο που θα έπρεπε να διαμετραματίσει προκειμένου να παράσχει πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Είναι αλήθεια ότι έχουν ένα ρόλο, αλλά ε, όπως αποδεικνύει η πρωτοβουλία της Γαλλικής Μη Κυβερνητική Οργάνωσης, οι ΜΚΟ γνωρίζουν και έχουν αποδείξει κατά τη διάρκεια όλη τη ιστορία τη Ευρώπη ότι το πράττουν και θα πρέπει να τις ενισχύσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Πολλές φορές είναι πιο επίμονες, πιο μαχητικές και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην τις, τους θέτουμε εμπόδια. Ναι, ε, πράγματι το Ινστιτούτο στο Βιλνίους έχει ένα ρόλο, αλλά πρόκειται για μια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό παίρνει χρόνο να κινητοποιηθεί. Ίσως οι ΜΚΟ να μπορούν να δραστηριοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ κυρία Σόγο. Ευχαριστώ. Ελέγχθησαν πολλά ενδιαφέροντα. Ε, θα είμαι και εγώ σε ίδιο μήκο Υπάρχει κάτι και ανάμεσα στη θέση της κυρίας Βιλόρ και της κυρίας Μπριγέρ. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ΕΛΚ και το Ινστιτούτο. Αυτό, αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Υπάρχουν δυνατά στοιχεία. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε πραγματικά, θα πρέπει να έχουμε προσώπους σε διαφορετικά επίπεδα. Ούτως ώστε να έχουμε την, ε, όλες τις ψυχές οι οποίες εκφράζονται. Λέγεται καμιά φορά ότι ε, η πολλή πολυμορφία δεν είναι κάτι καλό. Αυτό είναι λίγο παράξενο. Υπάρχει κάτι το οποίο ξεχάσαμε. Ε, η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης Εκεί δεν έχουμε περιορισμό αρμοδιοτήτων και είναι μια αρχή η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα για αυτόν τον αγώνα. Τώρα, σε αυτά που είπε η Βελό, θα μπορούσε κανείς να δει από μια άποψη ότι έχουμε πιλωτικά σχέδια. Υπάρχει μια εμπειρία, κάτι που ξεκίνησε σε μια χώρα μέλος και βλέπουμε μετά αν αυτό μπορεί να διευρυνθεί ε, φερπίν στη Γαλλία. Αυτό είναι το οποίο είναι το νόημα της ρήτρα. Δηλαδή, κάτι το οποίο φυσικά προσάπτουν συχνά όσον αφορά την πρόοδο την νομοθετική, πάντοτε είναι αυτό που ακούγεται τι θα γίνει στην πράξη, τι θα δώσει. Ναι, αλλά να, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε δει κάτι που ε, στην Ισπανία, εδώ και εκεί και βλέπουμε τι γίνεται στην πράξη. Αυτό μπορεί να συμπληρωθεί από κοινοτικά σχέδια, προγράμματα και να γίνει εκκίνηση κάποιων προγραμμάτων, να δούμε τι θα αποδώσουν. Δηλαδή πρέπει πράγματα να δούμε τι γίνεται στην πράξη για να διαπιστώσουμε αν μια ιδέα είναι καλή. Μόνο η πραγματικότητα μας αποδεικνύει το, το σωστό ή όχι μια ιδέα. Και κάτι τελευταίο. Ειλικρινά. Θα με ξέπλητε ότι στα, στατιστικές σε θέματα ε, ισότητας ανδρών ε, γυναικών ε, είναι αξιόπιστες σε, για τις 27 ε, χώρες. Λέγεται για συχνά ότι η στατιστική είναι μια, θα λέγαμε, ε, άλλη λέξη για το ψεύμα. Θα ήταν πραγματικά να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Τέλος. Όντως, ε, η, μια πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι πανάκια, αλλά θα σε ένα-δύο χρόνια ε, θα πρέπει ε, τα θεσμικά όργανα να προβληματιστούν, να δουν ποια είναι η πρόοδος σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας και να διαπιστώσει ενδεχομένως ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Και καταλήγουμε σε μια εποχή όπου πάρα πολλοί πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάθε άλλο παρά δημοκρατική. δεν, ε, δηλαδή, δηλαδή οι μηχανισμοί όσον αφορά δεν είναι μόνο προβληματικοί όσον αφορά την ισότητα ανδρών γυναικών. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Ε, σας ευχαριστώ. Διπανή, η κυρία Διπανή. Σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω κι εγώ ε, ανακατεμένα κάπως για να ευχαριστήσω Ναι, ε, ξέρω ότι υπάρχουν πολλές συνεδριάσεις ταυτόχρονα και καταλαβαίνω αυτό. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως να σας πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι που είμαστε εδώ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή σας που μας δέχτηκε και μπορέσαμε να εκφραστούμε. Είναι μια πρόοδος για τις γυναίκες να έχουν μια, ένα τέτοιο διάλογο. Τις προτάσεις της κυρία Μαρία Γκαμπριέλ σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σορών για μια ομάδα εργασίας σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, παίρνει χρόνο, είναι χρονοβόρα διαδικασία κάτι τέτοιο, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια τέτοια συνεργασία με την ομάδα εργασίας. Όσον αφορά το θέμα των στατιστικών, κυρία Σαρτιέ, ξέρατε Υπάρχει ένα βιβλίο που, που το θεωρώ ενδιαφέρον από τη στη Γαλλία δημοσιεύθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν στατιστικές για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. που δείχνουν πραγματικά ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα στο Βίνιους ε, καλά θα κάνει να συμπληρώσει το έργο του Ξέρουμε ότι ανάλογα ε, ντοκουμέντα υπάρχουν και στις χώρες μέλη. Καλό είναι να συμπληρωθούν, να υπάρξει μια συνέχεια. Είναι χρήσιμο θα έλεγα. Εγώ έχω μάθει πολλά πράγματα για, τους, για τα δικαιώματα των γυναικών. Και με τα μέτρα που ήδη έχουν εγκριθεί βλέπει κανείς ότι υπάρχει ήδη κάποια βελτίωση. Η κυρία Τόμσον τώρα. Άκουσα, αγωνίζεται πολύ για την παρουσία των γυναικών στο στην αγορά εργασία. Ξέρουμε είναι μια περίοδο κρίσεως και πραγματικά οι γυναίκες είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο ε, με την απασχόλησή τους, ε, τις, ε, όταν θα βγουν στη σύνταξη κτλ. ειλικρινά καταλαβαίνω ότι οι γυναίκες είναι σημαντικό να δουλέψουν και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουν την αναξαρτησία τους. Για την Λυπάμαι, δεν άκουσα το όνομα της εκπροσώπου της Επιτροπής. Α, ευχαριστώ που μου το λέτε. Ε, ε, όντως, εδώ έγινε πολύ μεγάλο έργο από τα θεσμικά όργανα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ε, υπάρχουν πολλά θέματα που εγώ δεν έχω αναπτύξει. Ε, υπάρχει κάτι το οποίο λάβαμε υπόψη. αντιμετωπίξαμε πολλά προβλήματα για να εντοπίσουμε το καλύτερο μοντέλο, να δούμε όλες τις νομοθεσίες. Έχουμε μικρά, μεγάλα κράτη, υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες. Προσπαθεί κανείς να έχει... Καμιά φορά τα σήματα είναι ανάλογα. Ε, για τη βία Φερπίν ε, είδαμε τι γίνεται στην Ισπανία. στην Ισπανία ε, οι στατιστικές που έχουμε ήταν ε, μια καταστροφή. Ε, έχουν γίνει, έχει γίνει πρόοδος όσον αφορά την προστασία των γυναικών, τα παιδιά, όλες αυτές οι πτυχές και σωστές, ε, σωστά μέτρα όπως η κατάρτιση του προσωπικού στην αστυνομία. Είναι πραγματικά μια πλήρη νομοθεσία που έχουμε εκεί αλλά έχουμε και άλλα μοντέλα δεν τα έχουμε ε, θα λέγαμε αξιολογήσει να πούμε τα υπέρ και τα κατά. Κάθε χώρα έχει μια νομοθεσία σε όλους τους τομείς και δεδομένα. υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία μπορούν να υπάρξει, μπορούμε να έχουμε μια ομοφωνία. Το μισθό για, την, για το γάμο Φερρυπίν εδώ πέρα έχουμε επιλέξει την Αυστρία. Γιατί θεωρούμε ότι καλύπτει καλύτερα τη γυναίκα. Κάτι που δεν ισχύει σε άλλες χώρες. Ε, έχουμε να κάνουμε δικαιώματα συγκεκριμένα. Τώρα, για την εκπροσώπηση σε πολιτικό επίπεδο η επιλογή μας ήταν η το Βέλιο, όπου τα δικαιώματα καταχειρώνονται σε συνταγματικά θα λέγαμε. Και επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε ότι κάνετε πολλά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι συνθήκες, οι οδηγίες. Αναφερθήκατε στην ε, ε, άδεια που μπορούν να έχουν οι γονείς, ε, πατρική ή μητρική. Τα θέματα της βίας. Μεγάλος είναι ο κατάλογος ο Ευρωπαίος πολίτης ξέρει τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει θέμα φυσικά ενημέρωσης. Αυτό που δεν έχει ο πολίτης είναι γνώση του τι ακριβώς γίνεται. Με αυτή τη ρήτρα προσπαθούμε να δείξουμε με αφορμή αυτό ότι υπάρχουν πρόοδοι σε όλους τομείς για τις γυναίκες με βάση τα υπάρχοντα μοντέλα όλα αυτά για να δείξουμε, με στόχο να δείξουμε ότι είναι σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να ε, επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον, ενδιαφέρον να δείξουμε τα μέσα που υπάρχουν, αλλά να ξέρουμε όταν εγκρίνεται ένα κείμενο, μια οδηγία, κάθε χώρα ανάλογα με το δικό της κοινωνικό μοντέλο και τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο το σύστημα, έχει επιπτώσεις έχει να κάνει αυτό, δηλαδή με ποιο μοντέλο μπορεί να επιλέξει κάθε χώρα, ανάλογα με τη δική της ε, κατάσταση και το δικό της σύστημα. Υπάρχουν διαφορετικές στάσεις, διαφορετικά κοινωνικά συστήματα. Ξέρουμε πραγματικά ότι είναι δύσκολο αυτό το έργο. Και δύσκολο να πετύχει κανείς μια συνένεση. Όντως όμως υπάρχουν πολλά μέσα. Η κυρία Μπόβαρ τώρα βλέπω έχει φύγει. Ε, πραγματικά εμείς δεν κρίνουμε τίποτα. Έχουμε μια αρχή ότι υπάρχουν διατάξεις σε, στη χέρια μας, σε διαφορετικά επίπεδα, όπως και στη διεθνή σύμβαση σε, σε διεθνές γραφείο εργασίας. Υπάρχουν επίσης τα, συστήματα, ε, τα εθνικά συστήματα προτασίας ε, μπορεί κανείς να βρει νομικές διατάξεις για... Έχουμε βρει διάφορες ρήτρε του πιο προνομίου κράτους. Προσπαθήσαμε με αυτή τη μελέτη να δούμε πώς με όλες αυτές τις διατάξεις διαφορετικές να καταλήξουμε σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά υπάρχει το θέμα των αρμοδιοτήτων. Ξέρουμε φυσικά ότι υπάρχουν όλες αυτές οι διάφορες αρχές. Παρόλα αυτά, θα σας τη δώσουμε αυτή τη μελέτη. Διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να δράσουμε σε διαφορετικούς τομείς προσπαθώντας να έχουμε ένα σφαιρικά ένα πρόγραμμα που θα μας οδηγήσει στο να καταλάβουμε σωστά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κάτι, να κάνουμε καλύτερα αυτό που κάνουμε, να είναι πιο ευανάγνωστο. Αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά υπάρχει το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να παρέμβουμε όπως ε, στα εθνικά δικαιώματα. Σίγουρα υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Κι αν γίνει συνταχθεί αυτή, συστηθεί συγγνώμη ομάδα εργασίας να το δούμε τότε. Προ... Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν κλείνοντας ίσως η κυρία Βεγλό μου έχει ζητήσει το λόγο συμπληρωματικά και έχω και κάποιε ερωτήσει που έχουν τεθεί, ίσως επίση και κάποιοι συνάδελφοι τώρα να θέλουν να πρόσθετε διευκρίνηση. Κύριε Αβεγλό, Διαπίστωσα ότι ξέχασα να απαντήσω σε ένα ερώτημα που μου θέσατε και επανέρχομαι. Είναι αυτό που ανέφερε η κυρία Σότ. Είναι πάντα δύσκολο να γνωρίζουμε τι είναι το βέλτιστο, τι είναι το καλύτερο. Και αναφερθήκατε στο δικαίωμα των, της διατροφής, του διαζυγίου και της διατροφής των παιδιών της διεκδίκησης ε, παιδιών μετά από διαζύγιο. Νομίζω ότι εδώ είναι ένα καλό παράδειγμα που μας δείχνει ότι υπάρχει λύση γιατί είναι δύσκολο κανείς να επιλέξει ποια είναι η βέλτιστη πρακτική στη διατροφή ή στο διαζύγιο γιατί οποιοδήποτε μέτρο και να πάρει κανείς εφαρμόζεται σε διαφορετικό πλαίσιο. Το εθνικό πλαίσιο Όπω ανέφεραν και οι συνάδελφοί μου, είναι πολύ διαφορετικό και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Ε, είναι ε, καλά παραδείγματα η διατροφή και το διαζύγιο. Για παράδειγμα, αν σε μια χώρα στην οποία υπάρχει πραγματική ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, εκεί δεν τίθεται καν ζήτημα διατροφή, Εκεί μπορεί να υπάρχει από κοινού γονική μέρημνα για το παιδί μετά το διαζύγιο. Αν όμω μιλάμε για μια χώρα στην οποία υφίστανται μεγάλες και σημαντικές διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων, Εκεί η διατροφή θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να βοηθά κατά κύριο λόγο τη μητέρα, γιατί διαφορετικά η μητέρα θα υφίσταται διακρίσεις, θα βρεθεί σε δυσμενή θέση. Άρα, σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και να σκεφτούμε γιατί είναι δύσκολο να βρούμε τη βέλτιστη πρακτική. Ο λόγος είναι επειδή δεν μπορούμε συστηματικά να προβάλλουμε το μοντέλο σε μια, μια, της χώρας μας ή μιας χώρας σε άλλες χώρες. Άρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το εθνικό πλαίσιο και το εθνικό νομικό σύστημα σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Ωραία, η κυρία Τόμψον είχε ζητήσει να επανέλθει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και που μου δίνετε την ευκαιρία να δευτερολογήσω. Είναι για τον, την καθηγήτρια την κυρία Βέρλο. Αναφερθήκατε στο Ινστιτούτο, στο Βίλνιους. Έχουμε μια θέση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάθε χώρα, κάθε κράτος μέλος πρέπει να δημιουργήσει ένα Ινστιτούτο για την, για την ισότητα των δύο φύλων. Όλες οι χώρες, εκτός από την Ισπανία έχουν εντάξει το Ινστιτούτο ή την Φορέα για την Ισότητα των Δύο Φύλων σε άλλους φορείς που έχουν σχέση για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα ή κάποιον άλλο τομέα των διακρίσεων. Και ε, θεωρώ ότι εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε επιδιώξει να μην εμπλέκεται, να, να, να, να, να γίνεται η διάκριση μεταξύ των διακρίσεων που οφείλεται στην ανισότητα των δύο φύλων και άλλες διακρίσεις όπως για παράδειγμα τις διακρίσεις κατά των μειονότητων. Οι γυναίκες δεν είναι μειονότητα, είναι ε, το 52% του πληθυσμού. Άρα θεωρώ ότι είναι προβληματικό να μπλέκουμε αυτά τα δύο ζητήματα, τι διακρίσεις κατά των μειονοτήτων και την ανισότητα των δύο φύλων. Θα ήθελα να ακούσω τις δικέ σα απόψει από αυτού. Το θεωρώ επίση σημαντικό γιατί η Επιτροπή για τα ενισότητα των δύο φύλων εδώ στο Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να εφαρμόσει μια αξιολόγηση. Πρώτα απ' όλα θα εξετάσουμε κατά πόσο δημιουργήθηκαν αυτοί οι φορεί και μετά, αυτή στιγμή δημιουργήθηκαν, θα εξετάσουμε τη λειτουργία του και πόσο αποτελεσματική είναι. Θα ήθελα να ακούσω τι απόψει για αυτό το ζήτημα. Και μια... και μια ερώτηση προς την ίδια κατεύθυνση. Αυτό που ρώτησε η κυρία Τόμσεν, υπάρχουν αυτά τα Ινστιτούτα, τα Ιδρύματα και τα Παρατηρητήρια. Ποιο είναι ακριβώς το έργο τους, πώς λειτουργούν, τι παράγουν, ποιο είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος που προκαλούν και πώς αξιολογούνται οι δημόσιες πολιτικές. Το ερώτημα αυτό έχει τεθεί. Οι εμπειρογνώμονές μας δεν απήντησαν αποτίμηση κρατικών πολιτικών είναι καθοριστική σημασίας για μας. Γιατί πώς να μπορέσουμε εμείς να δώσουμε την εντύπωση ότι μια ή άλλη ρήτρα την χάνει καλύτερης αντιμετώπισης ε, σε μια χώρα, οπότε να προωθήσουμε κατά συνέπεια και ένα μοντέλο, εάν δεν είναι ε, και δεν ξέρουμε πώ αποτιμώνται οι κρατικέ πολιτικέ. Νομίζω και οι δύο παρατηρήσει τη κυρία Τόμψον και οι δικέ μου είναι... συγκλίνουν. Θα ήθελα λοιπόν ε, στι απαντήσει σα να λάβετε υπόψη τι δύο αυτέ διαστάσει. Κατά πρώτον, να πω σε όλους ότι είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνει κανείς τέτοια θεσμικά στοιχεία και τις εξελίξεις στα διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσπαθήσαμε στο πρόγραμμα Queen, αλλά Κάτι που ισχύεται μία εβδομάδα μετά μπορεί να αλλάζει. Ο καθένας στην κάθε χώρα ξέρει ότι ο χώρος αυτός εξελίσσεται πολύ δυναμικά. η θέση της ισότητας των, της φίλων σε αυτούς τους θεσμικούς φορείς ήταν κάτι που το έχουν αναφέρει πολλοί συνάδελφοι από την Ουγγαρία, την Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκείνοι χαρτογραφούν το βαθμό στον οποίο οι θεσμικοί μηχανισμοί έχουν ενοποιηθεί και κοιτάνε ποια μοτίβα προκύπτουν από, αυτά, από αυτούς τους συνδυασμούς ε, τι γίνεται με τους διαφορετικούς φορείς της αντιμετώπισης διακριτικής μεταχείρισης κατά των γυναικών, τους συμβουλευτικούς φορείς. Βλέπουν που υπάρχει ο μεγαλύτερος βαθμός σύγκλησης ε, στους φορείς αντιμετώπισης της διακριτικής μεταχείρισης η διακριτική μεταχείριση όταν αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα σε όλους τους τομείς ε, αντιμετωπίζεται και αποτελεσματικότερα. Τώρα, όταν ε, μιλάμε για συμβουλευτικούς φορείς, όταν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, βλέπουμε ότι επίσης υπάρχει και λιγότερη ενοποίηση. Τέλος πάντων, ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα δυναμικός και το βιβλίο αυτό μόλις δημοσιεύτηκε, είναι πολύ πρόσφατο, οπότε δίνει μια επισκόπηση του βαθμού στον οποίο συμβαίνουν όλα αυτά βρήκαμε ότι σε χώρες όπως την Πορτογαλία έχουμε αυτή τη στιγμή μια τρόποντινά βέλτιστη πρακτική. Μια μορφή συνεργασίας που είναι αποτελεσματική. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα και αυτό είναι η δική μου καλύτερη πρόβλεψη για το τι μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά ως μορφή. Διότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες για την ισότητα των φύλων στον τομέα αυτό αλλά αν δεν θέλετε να εργάζονται αυτοί προς όφελος της ε, ετεροσεξουαλικής με, με ανώτερης τάξης και με υψηλή μόρφωση γυναίκας, θα πρέπει να το φροντίσουμε αυτό. Υπάρχουν γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες και δεν καλύπτονται. Χρειάζονται λοιπόν πολιτικέ ισότητα των φύλων που να καλύπτουν τι ανάγκε και τα δικαιώματα και αυτών, όλων των γυναικών. Η ρήτρα δείχνει πολλές φορές ε, τι συμβαίνει σε αντίθετες περιπτώσεις, όπως στην Αυστρία με το γάμο ή στην Ισπανία, όπου δίδεται η δυνατότητα του γάμου μεταξύ ομοφιλόφιλων ζευγαριών. Στην Αυστρία όμως είχα πολύ καλύτερα παραδείγματα, διότι είχα εργασία μερικής απασχόλησης. Αλλά υπάρχει πρόβλεψη για το συνδυασμό της εργασίας και του κοινωνικού βίου εκεί. Η αρχή της ρήτρα που θα έπρεπε να δούμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, να σκεφτούμε δηλαδή ως ένα εργαστήρι παραγωγή δημιουργικών ιδεών και συζήτηση για το τι είναι το καλύτερο, είναι ένα πρώτο βήμα και μετά να προχωρήσουμε. Ελπίζω να απάντησα. Όχι, όχι, ρωτήσατε και για το. Ναι, μίλησα για την αποτίμηση των δημοσίων πολιτικών. Ναι. Απλώ δεν ήμουν βέβαιο ότι κατάλαβα καλά. Να προσθέσω κάτι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Σε σχέση με όλα αυτά. Και τη ρήτρα για την πλέον ευνοημένη Ευρωπαία. Πρέπει να κοιτάξουμε να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις. Διότι έγραψε ένα βιβλίο το 2005 για τις γυναίκες στην Ευρώπη και κατέληξα ότι τις καλύτερες επιδόσεις στην ιεραρχία, στην αγορά εργασία την έχει η Πορτογαλία. Εγώ είμαι Δανέζα. Ε, νομίζω ο αριθμό για μα είναι 23%, για τη Γερμανία 26%. Όμω, η άποψη που έχουμε για την Πορτογαλία γενικώ στην Ευρώπη είναι ότι είναι φτωχέ οι Πορτογαλίδες και όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έχει πολύ καλέ επιδόσει από την πραγματικότητα. Έχει πολύ καλέ επιδόσει η Πορτογαλία. Σα ευχαριστούμε που υπογραμμίσατε το στοιχείο αυτό. Κυρία Βερλό, θέλετε να συμπληρώσετε. Ναι, όπως και για τη ρήτρα. Ξέρουμε ότι στον τομέα της βίας η Αυστρία και η Ισπανία έχουν λάβει πολύ καλά μέτρα. Όχι οι σκανδιναβικές χώρες, όχι η Ολλανδία, όχι η συνήθιση υπόπτη. Παρομοίως, καλές πρακτικές υπάρχουν στη Σλοβενία. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην παραμένουμε στα στερεότυπα. ως προς την αποτίμηση των δημοσίων πολιτικών και όπως το ζήτησε η Πρόεδρος, για το mainstreaming των φίλων ε, νομίζω ότι για τέτοιους σκοπούς είναι χρήσιμο αλλά έχουμε χάσει κάπως την έννοια της μελέτης αντικτύπου χρειάζονται και παραδείγματα από την ιστορική εξέλιξη για να εντοπίσει κανείς μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα, γιατί κάποια πράγματα δεν ισχύουν πλέον. Για τα παραδείγματα θα το δούμε στα συμπεράσματα. Κυρία Ντουπανή. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. να μιλήσω για τα μοντέλα κάποιων χωρών που γνωρίζουν, γνωρίζω καλά. Για το γάμο, αυτό που λέτε είναι όντως σημαντικό, διότι επιλέξαμε το παράδειγμα της Αυστρίας αλλά και της Ισπανίας, που δίνει τη δυνατότητα και στους ομοφιλόφιλους να παντρευτούν. Λόγω χάρη, στις μικρές χώρες μου φαίνεται σημαντικό να δούμε τι γίνεται. Να δώσω κάποια παραδείγματα όπως για την ε, γονεϊκή ευθύνη στην Εστονία. Στην Εστονία ορίζεται η γονεϊκή μέρημνα ανάλογα με την οικογενειακή σχέση ή σε άλλες χώρες ανάλογα με το σεξουαλικό προσανατολισμό και επιλογές. Στην Λιθουανία επίσης υπάρχει το θέμα της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας αλλά και στο νόμο για την ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ε, χαρτογράφηση, όπως είπα, έπρεπε να αναδείξει και τις ελλείψεις ισορροπίας Κάποιες χώρες που τι έχουμε ήδη ξεχωρίσει για κάποιο συγκεκριμένο τομέα δεν τι αναφέρουμε και δεύτερη φορά. Για κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες λοιπόν ε, ας είναι βέβαιο ότι δεν τις, ε, η αποσκόπηση δεν σημαίνει ότι τις αναφέρουμε αρνητικά. Τώρα για την αποτίμηση των πρακτικών Είναι πολύ σημαντικό παρόλο που δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ιδίω από την άποψη του προπολογισμού, όπω διαμορφώνεται σήμερα, θα πρέπει να τα σκεφτούμε. Κοιτάξτε, με είδη συμπεράσματο, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή μα, να ε, συνοψίσω κάποιε ιδέε και κάποιου γενικού προσανατολισμού. Το πρώτο στοιχείο που με φαίνεται σημαντικό και όπου πιστεύω ότι υπήρξε συμφωνία είναι ποια είναι η φιλοσοφία μας στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι η νομιμότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο. Η ισότητα ενώπιον του νόμου. Δηλαδή όχι η ευνοϊκή μεταχείριση μιας μερίδας του πληθυσμού έναντι κάποιας άλλης, αλλά η ίση κατάσταση όλων ενώπιον του νόμου. Ποια φιλοσοφία λοιπόν διέπει το έργο μας. Ο καθηγητής Σορών μας το είπε και νομίζω ότι είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη ως γυναίκες και άνδρες πολιτικοί αναζητούμε να δώσουμε ένα ανθρωπινότερο πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια θετική ένωση. Στην πράξη συνειδητοποιώ ότι αυτό τον ανθρώπινο χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον δίνουν στην πραγματικότητα οι πολίτες. Αυτά ως προς τη φιλοσοφία μας. Τώρα για τις ημερομηνίε. Δύο ημερομηνίε είναι σημαντικές. 2020. Όλοι οι στόχοι σύγκλησης, όλοι οι στόχοι της Ευρώπης το 2020 αντικατοπτρίζονται σε όλα τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Η θέση των γυναικών στο χώρο εργασία. Η μισθολογική ισότητα. Η θέση ανδρών και γυναικών στην κοινωνία. βλέπουμε στόχους πολύ σαφώς ε, καθορισμένους από πολιτικής άποψης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την προοπτική του 2020. Υπάρχει συνένεση σε αυτό το σημείο. Η δεύτερη ημερομηνία στην οποία δοθήκε έμφαση σήμερα μέσα από τις συζητήσεις μας είναι το 2014. Το 2014 οι ευρωεκλογές και η ανανέωση του σώματος του Ευρωκοινοβουλίου καθώς και του σώματος των Επιτρόπων όπως το θύμισε ο καθηγητής Σωρών είναι καθοριστική σημασία. Θα υπάρχει εκεί και ένας, πολιτικός, ένας νέος πολιτικός προσανατολισμός. Είναι ένα στάδιο, ένα ορόσημο το 2014. Ήθελα λοιπόν να δούμε ε, συνδυασμένα και σε μια κοινή προοπτική αυτές τις δύο ημερομηνίες, 2014-2020. Κάτι άλλο που υπογραμμίστηκε είναι η ποικιλομορφία των νοοτροπιών, η διαφορετικότητα των εθνικών πολιτικών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, Υπάρχουν εργαλεία για να καλυφθεί αυτή η διαφορετικότητα, όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτή τη διαφορετικότητα, την κοινωνική, την ε, ποικιλομορφία στις νοοτροπίες. Οποιαδήποτε ταξινόμηση φαίνεται τεχνητή, επίπλαστη. Οποιαδήποτε οριζόντια ε, ταξινόμηση, όπως θύμισε τώρα η, ε, η κυρία Τόμψεν, ε, μπορεί να στέκεται στο ένα ή το άλλο σημείο κάποιες εμπειρίες από ένα συγκεκριμένο κράτος που μπορεί να είναι θετικότερες από ένα άλλο. Το άλλο σημείο, δύο ακόμα σημεία στα οποία θέλω να σταθώ, είναι ότι δεν υπάρχει από ιστορικής πλευράς γραμμική πρόοδος για το θέμα αυτό. Για την ισότητα των πολιτών τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, την ισότητα ανδρών γυναικών υπάρχει ε, αυταπάτη αν πιστεύουμε ότι υπάρχει συνεχής και γραμμική πρόοδος. Είμαι ιστορικός ειδικευμένη στην ιστορία των γυναικών και σας διαβεβαιώ. Σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους οι γυναίκες στην αρχαιότητα λόγω χάρη είχαν εξαιρετικά σημαντικές ε, θέσεις ή στο Μεσαίωνα ή στον 18ο αιώνα. Στις περιόδους αυτές όπου κατέλαβαν στην κοινωνία σημαντικές θέσεις, ε, ε, στις περιόδους αυτές ε, πολλές φορές ακολουθού, από τις περιόδους αυτές ακολουθούσαν άλλες όπου υποβαθμίζονταν οι γυναίκες. Για τις ευρωπαϊκές λοιπόν πολιτικές των οποίων ηγούμαστε για το έργο του Ιδρύματος ε, Ισότητας των Φίλων στο Βίλνιους πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Διότι δεν ονειρευτήκαμε, δεν φανταστήκαμε ότι είμαστε οι πρώτοι και οι καλύτεροι ή οι τελευταίοι και οι τελειότεροι στην οικοδόμηση της ισότητας των φύλων για την Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ταπεινοί και πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για ένα έργο διαρκές, συνεχιζόμενο. Η κοινωνία συνεχώς μεταβάλλεται υπάρχουν σοβαροί τριγμοί, μιλήσαμε για την κρίση λόγου χάρη, και αυτοί οι σοβαροί κλειδονισμοί κάποιες φορές μας οδηγούν να μας φέρουν αντιμέτωπους με την πραγματικότητα. Ιδού Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τις τις εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν σήμερα, τις συναδέλφους βουλευτές που κινητοποιήθηκαν και νομίζω Πρόεδρε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και για πολύ καιρό κιόλας επί του θέματος. Ευχαριστώ όλους και όλες που ήρθατε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς μας που διευκόλυναν την επικοινωνία μας. Και ως προς το στόχο αυτό θα κάνουμε πολλά ακόμα πιστεύω στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε.